So, dear um, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε αργήσει 7 λεπτά γιατί ξεκινήσαμε από τις 9 το πρωί μαζί με την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Επομένω, στην ώρα μας είμαστε, απλώς συνεχίζουμε. Είχαμε, θα, είχαμε μια καλή και επικοδομητική συζήτηση για τα πολιτιστικά προϊόντα και τον έλεγχο των εισαγωγών. Τώρα όμως Περνάμε στην ε, συνεδρίαση καθαρά της δικής μας Επιτροπής Εθνούς Εμπορίου. Ναι, το σημείο 2 καταρχάς στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης και ρωτώ αν έχετε κάποια πρόταση για τροποποίηση. Αν όχι εγκρίνεται. Σημείο 3. Πρακτικά. Ως ήθιστε Τα πρακτικά κρίνεται ότι εγκρίθηκαν εάν δεν έχουν ε, αντιτεθεί παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης. Σημείο 4. Αποφάσεις των συντονιστών. Σας έχουν κοινοποιηθεί σχεδόν τα ίδια με αυτά που συμβαίνουν και στα πρακτικά και για τα πρακτικά. Άλλες ανακοινώσεις, από πλευράς μου τώρα. Ως ήθιστε έχουμε μετάδοση από το διαδίκτυο. Γι' αυτό να μιλάτε καθαρά στα μικρόφωνα. Να ξέρετε ότι μπορεί να σας δει ολόκληρος ο κόσμος. Εκατομμύρια πολιτών. Ναι, σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε. από το Ελσίνκι στην Θεσσαλονίκη και από τη Λισαβόνα στο Λίμπουργ. Καλώς ήρθατε την κυρία Κάτταενεν της Άλντε που διαδέχεται τον κύριο Τάκουλα από τη Φιλανδία. Αν δεν απατώμε, καλώς ήρθατε και καλή δουλειά στην... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΕΝΦ. Η ΕΝΦ όρισαν την κυρία Φράντς Ζαμί ως συντονίστρια. Παίρνω στο σημείο 6. Μέλλον τροφίμων και γεωργίας. Με την εξή δυσκολία. Ότι ο εισηγητής αυτού του υπέροχου θέματος λείπει. Ο κύριος Κέλλη. Έχει το ΕΛΚ να μας υποδείξει γιατί αγνοείται. Πού βρίσκεται. Καλά, λοιπόν, πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Άγκρη που έχει την κατουσία αρμοδιότητα για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Η Επιτροπή λοιπόν Γεωργίας προτίθεται να διατυπώσει ιδέες που θα απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις λάβει υπόψη της αυτή όταν ετοιμάσει την, τις νέες προτάσεις για την κοινή πολιτική. Και δεν θα αργήσει αυτό. Στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα προκύψει και αυτή η πρόταση. Αναμένεται η Επιτροπή να καταθέσει σχετικά σύντομα προτάσεις κάπου στο τέλη Μαΐου Ας αρχίσουμε όμως. Και ας δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Να μας εξηγήσετε παρακαλώ πώς έχετε σχεδιάσει την ε, ε, μεταρρύθμιση, τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε κτλ. Παρακαλώ. Thank you, I'll be, I'll be very brief, uh, as you... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όπως είπατε πολύ σωστά, προβλέπουμε να υποβάλουμε τις νομοθετικές προτάσεις κάπου στα τέλη Μαΐου λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο οι οποίες φυσικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του αντικειμένου και του μέλλοντος ε, της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα όσον αφορά την επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, αλλά Θέλω να σας πω ότι επιχειρούμε να έχουμε μια μεταρρύθμιση εξυγχρονισμού εντάσσοντας περισσότερο τους στόχους ε, της κλιματικής αλλαγής και τους βιώσιμους στόχους ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας. Μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα διασφαλίζει ότι η οικονομική στήριξη θα πηγαίνει στους αγρότες που δεν χρειάζονται περισσότερο και με πιο ισότιμο τρόπο. Μια ΚΑΠ η οποία θα αξιοποιεί την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία ώστε να βελτιώνει την βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η βασική στόχη τη επόμενη ε, επερχόμενη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Έχω δύο παρατηρήσει, κύριε Πρόεδρε, για το σχέδιο γνωμοδότηση. Να περιμένω ενδεχομένω ε, μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση τη Επιτροπής πριν σας παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κανένα δυο στοιχεία για τις απόψεις της Κομισιόν σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και το Διεθνές Σύστημα Εμπορίας. Ειδικότερα ε, όσον αφορά τις συζητήσεις για το πρασίνισμα στον ΠΟΕ και το ζήτημα που έχουμε γενικότερα με τις ΗΠΑ. Τρία είναι ζητήματα, τα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, που θεωρούμε ότι δημιουργούν ε, τη σύνδεση μεταξύ του Διεθνούς Θεματολογίου για το εμπόριο και του περιεχομένου της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα στην επόμενη ΚΑΠ θα διατηρήσουμε την, ε, τον προσανατολισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής προς την αγορά ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τροφίμων και της γεωργίας της Ευρώπης. Καλό θα ήταν, πιστεύω, η γνωμοδότηση να ενθαρρύνει ε, τη συνέχιση αυτής της ε, κατεύθυνσης του προσανατολισμού της γεωργικής πολιτικής προς την αγορά. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, και αυτό αφορά το περιεχόμενο και τη δομή της επόμενης ε, γεωργικής πολιτικής, παρότι η μεγαλύτερη παρουσία στις διεθνείς αγορές είναι κάτι καλό. Αυτό αναγνωρίζεται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γεωργία στην Ευρώπη εκτίθενται σε μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών ε, διότι είναι εκτεθειμένοι σε διεθνείς αγορές. Συγγνώμη, εκτίθενται σε μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών και αυτό ε, επηρεάζει τα εισοδήματα των Ευρωπαίων αγροτών. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι στην επόμενη εκδοχή της ε, ΚΑΠΑ ε, θα υπάρχουν μέτρα που θα βοηθούν τους γεωργούς σε δύσκολες εποχές. Θα τους βοηθούν να επιβιώνουν τις εποχές μεγάλης αστάθειας και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα, στην επισήτηστική αλυσίδα. Πιστεύω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συζήτηση της παρουσίας Επιτροπής. Ε, το τρίτο που θέλω να πω κύριε Πρόεδρε είναι ότι το σχέδιο γνωμοδότησης στην παράγραφο 3 υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας, ότι προσθέτουν αξία. Εμείς θα θέλαμε να αναφέρετε και κάποια αναγνώριση ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες της επιτυχίας μας στις υπερπόντες αγορές όσον αφορά τα τρόφιμα είναι ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα έχουν πολύ καλή φήμη όσον αφορά την ποιότητα, την διατροφική αξία και τους τρόπους παραγωγής ε, λόγω των υψηλών πρότυπων ε, καλής μεταχείρισης των ζώων και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Η τήρηση όλων αυτών των πολύ υψηλών πρότυπων και απαιτήσεων ε, συνεπάγονται πολύ σημαντικά υψηλά κόστη για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό στο μέλλον, όπως ήταν και στο παρελθόν, να παρέχουμε επαρκές επίπεδο ε, υποστήριξης εισοδήματος για τους Ευρωπαίους αγρότες, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν ε, τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τα υψηλότερα ε, πρότυπα, ώστε να ξεχωρίζουν στις διεθνείς αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρίστερο Ρόβολτ θα αντικαταστήσει τον κύριο Κέλλη. Τι δίνω το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σας συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου μας, ο δεν μπορέσε να έρθει. Σα διαβάζω το κείμενό του. Δεν, είναι, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη με το θέμα. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη δυνατότητα της αξιολόγησης ε, της κατάστασης του ευρωπαϊκού Πληρωτικού τομέα και της συμβολής του στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, θα ήθελα να εγείρω κάποια σημεία εδώ τα οποία καταγράφονται στο σχέδιο γνώμοδο της Επιτροπής μας. Καταρχάς, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην ολοκλήρωση των στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής και κυρίως στην εξασφάλιση ε, ισότιμων συνθήκων και αξιοπρεπών συνθήκων επιβίωσης και διαβίωσης των ε, γεωργών αλλά και προϊόντων ε, ικανοποιητικής πυρότητας για τον καταναλωτή. Επίσης θέλαμε να επισημάνουμε ότι το τομέα τροφίμων και γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο στις εξαγωγές καθώς ε, οι αγορές εκτός Ευρώπης παίρνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Είναι τεράστιος ο ρόλος ε, των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στις εμπορικές συναλλαγές και τις τωρινές διαπραγματεύσεις μεταξύ, με διάφορες ε, χώρες. Ο σημαντικός ρόλος της γεωργίας και στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων για διμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες αλλά και πολυμερές επίπεδο, που δείχνει ότι οι κανόνες, είτε τη φυτοϊγιεινή, είτε της γεωγραφικής προέλευσης, είτε της ευημερία των ζώων, οι προδιαγραφές ε, και οι απλουστευμένες διαδικασίες έχουν τεράστια σημασία και πρέπει να διαφυλαχτούν. Καλώς ορίζω την πρόοδο που επετεύχθη στην προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των πρόσφατων δημερών ε, διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων ε, και τροφίμων και κυρίως της προστασίας γεωγραφικής προελεύσεως σε ε, τρίτες χώρες. Ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Ωστόσο, ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μεριμνήσουμε και θα υποστηρίξουμε το γεωργικό μας τομέα. Γι' αυτό και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των ελληνών αλλά και μελλοντικών ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες να προχωρεί με μέγιστη φροντίδα και προσοχή σε μέτρα απελευθέρωσης τομέων σχετικών με τη γεωργία και τα τρόφιμα, με μεταβατικές διατάξεις, με διασφαλιστικές δικλίδες και με αποκλεισμό από την ε, απελευθέρωση των πιο ευαίσθητων προϊόντων. Ο γεωργικός τομέας ιδιαίτερος θα μπορούσε να αφορά ε, στην προκειμένη περίπτωση ε, δημητριακά, ζάχαρη γαλακτοκομικά, ε, βόηο κρέας και άλλα αντίστοιχα είδη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για την υποστήριξη και σε επίπεδο της υπολογική του ΠΟΕ των ε, εγχώριων προϊόντων, κάθε μέτρο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, καλό τους εμπορικούς εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευθούν ώστε να σταματήσουν τις εγχώριες ενισχύσεις και τα μέλη της ΠΟΕ που εξακολουθούν να επιβάλλουν ενισχύσεις στις εξαγωγές καλούνται να υλοποιήσουν την υπουργική διακήρυξη για τον ανταγωνισμό σε εξαγωγές ε, του Ναϊρόμπι του 2015 και επίσης καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να προστατέψουμε τις να στηρίξουμε τις αμυντικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση σε σχέση με εφιστάμενους και ε, περχόμενους φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές ε, και στην πρόσβαση σε τρίτες αγορές, ιδιαίτερα στο χωρέα των τροφίμων και, των, ε, και της γεωργίας. Αυτό έχει να κάνει με τη συμφωνία εταιρική σχέσης και την πρόσβαση σε αγορές. Καλώ τους αδέλφους λοιπόν να έρθουν σε επαφή μαζί μου εν ευθέτω χρόνο για να διαμορφώσουμε το κείμενο της νομοδότησης. Αυτά λέει ο κύριος Σον Κέλλη και τον ευχαριστούμε. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, μια σύντομη παρατήρηση προσωπική, έχοντας παρακολουθήσει επί χρόνια την εμπορική πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε το γεωργικό τμήμα των διαπραγματεύσεων. Έχει να κάνει ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο με μικρά ποσά μεν, αλλά με έχει τεράστια απήχηση στην κοινή γνώμη και αντίκτοπο αν ληφθούν αρνητικές αποφάσεις. Γι' αυτό και απευθύνω δραματική έκκληση χωρίς να είμαι μέλο τη Επιτροπή Γεωργίας. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει και για την επικοινωνιακή πολιτική με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβανομένων υπόψη και των διαφορών ευαισθησιών που αισθάνεται ο Ευρωπαίος πολίτης. Ευχαριστώ. Σαφές το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Η Καρολίνη είναι ε, εδώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον κύριο Ερίκα Αντριέου, είναι ο σκιώδης εισηγητής, αλλά είναι σε άλλη επιτροπή και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Καταρχάς, For opinion. Ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη για την γνωμοδότηση αυτή. Ε, συνάδει με το πνεύμα της επι... ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να αλλάξει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ, ε, οι οποίες ε, από τη δεκαετία του 90 κατευθύνονται κυρίως προς τις εξωτερικές αγοράς. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία για την χρηματοδότηση στο σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής. Καταρχάς, ο κοινός κανόνας της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ε, της ασφάλειας τροφίμων, ε, του περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της μελλοντική ε, ΚΑΠ. Θα πρέπει να σταματήσουμε να υποδαβλίζουμε την ε, ε, γεωργική μας πολιτική μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών και μετά να δίνουμε ενισχύσεις στους γεωργούς για να υποστηρίζουν το εισόδημά τους. Ε, βρισκόμαστε σε περίοδο περιορισμών στον προπολογισμό και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί προ τον εαυτό μα. Η γεωργία δεν θα πρέπει να είναι μια μεταβλητή στι διαπραγματεύσει. Η γεωργία δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν σαν όλα τα υπόλοιπα. Δεσμεύει τη γη μα, τα τρόφιμά μα, την ανθρώπινη υγεία. Και γι' αυτό ακριβώ είναι επιλογή τη κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μάχη για τους πιο ευάλωτους τομείς ε, και να υπάρχει ένας κατάλληλος ε, επίπεδο προστασίας ε, συμπεριλαμβάνοντας τα πιο ευαίσθητα προϊόντα από τις, και να αποκλείονται στις εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να Ευνοούμε το εμπόριο το οποίο θα βασίζεται σε κοινωνικά πρότυπα, σε περιβαλλοντικά, σε πρότυπα υγεία ε, και ευημερία των ζώων. Επίση, πρέπει να υπάρχει καλύτερη χνηλασιμότητα των προϊόντων που εισάγουμε. Το 2018 υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα υγεία τα οποία αυξάνονται και πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για του πολίτε μα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να γνωρίζουν τι τρώνε. Και τέλος, θα πρέπει να σταματήσει η ενίσχυση να είναι πρόβλημα για τις ε, εξωτερικές σχέσεις. Πρέπει να είναι μία από τις λύσεις. Λέγεται ότι δεν είναι ε, οι εμπορικοί κανόνες ευνοϊκοί για τις χώρες του Νότου και ευνοούν ε, την ανάπτυξη άλλων περιοχών του κόσμου και πιέζουν κυρίως τους γεωργούς να μεταναστεύσουν σε πιο έφορη γη. Θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε την κοινή γεωργική πολιτική μας και την εμπορική πολιτική μας και θα πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των χωρών του Νότου, ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν αυτονομία σε θέματα τροφίμων και να μπορέσουν να μην ε, καταφεύγουν σε μετανάστευση και να ε, ε, μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Δεν θα πρέπει η γεωργική πολιτική και η εμπορική πολιτική να είναι μία εναντίον ε, τη άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το μέλλον του ευρωπαϊκού προγράμματος της μου ε, για την ανθρωπιότητα στο σύνολό τη, ε, διακυβεύεται σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η ομάδα του ECR μπορεί να υποστηρίξει τη γνωμοδότηση και τις θέσεις που εκφράζει ο συντάκτης. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να άρουμε τους εμπορικούς φραγμούς και να υπάρχει πρόσβαση σε τρίτες αγορές. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση είναι να δημιουργηθούν νέοι φραγμοί. Γνωρίζουμε ότι περισσότεροι επηρεάζουν τα γεωργικά προϊόντα και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα την απελευθέρωση των αγορών, κυρίως για τα πιο ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα και να δούμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν ε, ποσοστώσεις, ε, δασμοί, μεταβατικές περίοδοι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ίσως και κάποιες ε, ρήτρε διασφάλισης και να εξαιρούνται τα πιο ευαίσθητα προϊόντα από το εμπόριο. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια καθολική προσέγγιση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ατομικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πρέπει να εξετάσουμε και κάποιους περιορισμούς. Η ΚΑΠ είναι μία από τις πιο σημαντικές κοινέ πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να εξετάζεται εκτός πλαισίου ε, και ξεχωριστά από το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εξετάσουμε και τι γίνεται με την επανεθνικοποίηση, να δούμε και τα στοιχεία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Και αυτό ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγγυάται η κοινή πολιτική. Πολύ συχνά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γίνεται λόγος για την τοπική πραγματικότητα, την κατάσταση που ισχύει, τις τοπικές συνθήκες της γεωργίας και θα πρέπει να έχουμε κατά νου την ποικιλομορφία της γεωργίας, την ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής, να εξετάσουμε κλιματολογικές συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες ε, και περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ευαισθητοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία συγκεκριμένη ερώτηση τώρα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία ε, πρέπει να ληφθούν. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε το θέμα σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται καλούς ε, κανόνες σε νομικό επίπεδο που μας επιτρέπει να ε, μπορούμε να προωθήσουμε τους κοινού στόχους που έχουμε θέσει και βάσει και των ευρωπαϊκών συνθήκων. Ταυτόχρονα ε, μπορούμε να τηρούμε και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι διεθνείς δεσμεύσεις να λαμβάνουν υπόψη τους και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Να δώσω για πρώτη φορά το λόγο στην κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά και καινούργια εδώ στην Επιτροπή σας. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και σας ευχαριστώ και για το καλωσόρισμα. Όσον αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργία στην ενή αγορά, Υπάρχει όλο αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας και φυσικά και ε, να πληρούνται συγκεκριμένε περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι παγκόσμιες απαιτήσεις όσον αφορά την εμπορική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η ΚΑΠ πρέπει να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα κυρίως για την επιμερία των ζώων και για τη μικροβιακή εντοχή. και να υπάρχουν και ενδείξει ε, ε, προέλευση. Όταν αναφερόμαστε στο εμπόριο και στη γεωργία, ε, έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν ωφέλη για το ελεύθερο εμπόριο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να προστατεύσουμε κάποια στοιχεία στη γεωργία, στις εμπορικές μας συμφωνίες, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες ανοίγουν νέες αγορές για τα ευρωπαϊκά προϊόντα συνεχώς. εμπόριο με προσανατολισμό στις εξαγωγές θα προσφέρει τη δυνατότητα στους γεωργούς να υποφοληθούν αυτών των συμφωνιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού παγκοσμίω. Ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι οι ενισχύσει και οι κανόνες του ΠΟΕ. Καταργούν καταργήθηκαν όλες οι ενισχύσει στον Ναϊρόμπι το 2015 και θα πρέπει να ζητήσουμε το ίδιο και από τους εταίρους μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη γνωμοδότηση του κυρίου Κέλλη και τον ευχαριστώ για ένα πολύ ισορροπημένο ε, κείμενο. κύριος Μπούχνερ. Πράσινη. Ευχαριστώ και εγώ. Θεωρώ ότι είναι καλή η έκθεση του κυρίου Κέλλη ως πρώτη πρόταση και σημείο εκκίνησης. Θα ήθελα ωστόσο να προβώ κάποιες προσθήκες και παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη γεωργία και τη διατροφή του μέλλοντος. Δηλαδή, δεν ε, πρέπει να μας απασχολήσει μόνο το ο κέρδος και αναφέρομαι σε μια οικολογική, σε μια ε, ισοδίκαιη ε, γεωργία και για τους γεωργούς τους δικούς μας αλλά και για τις άλλες χώρες του κόσμου. Πρέπει να αποφύγουμε τις καταστροφικές συνέπειες της εμπορικής πολιτικής που έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα στο νότιο ημισφαίριο. Παράγουμε σε πολύ χαμηλές τιμές τρόφιμα, με πολύ δυσμενείς συνθήκες οι οποίες καταστρέφουν το περιβάλλον. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ε, τα προβλήματα που προξενεί στην κλιματική αλλαγή, στην ε, ε, εκπομπή μεθανίου, στην ενίσχυση των μεταφορικών ροών, στην απολία της βιοπικιλότητας ε, που έχει τεράστια ε, που έχει εμφανιστεί σε τεράστιες διαστάσεις λόγω της χρήσης των ζυζανιοκτώνων και πολλά άλλα προβλήματα και το γεγονός ότι είναι τόσο κρίσιμη κατάσταση αποδεικνύεται και από την ε, εμφάνιση ανθεκτικών στα αντιβιωτικά οργανισμών που προκαλούν στην Ευρώπη τεράστιο αριθμό θανάτων και μάλιστα τα αντιβιωτικά αυτά προέρχονται, αυτό αποδεικνύουν και οι εκθέσεις ε, των ειδικών, από την γεωργία. Με τον περιορισμό λοιπόν των εξαγωγών ε, των, ε, του κρέατος δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η γεωργική άλλωστε παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες ταλαιπωρείται και κινδυνεύει από τις ε, δικές μας εξαγωγές. Επομένως χρειάζεται μια προσαρμοσμένη, μια νέα πολιτική εμπορίου. Ε, έχω λοιπόν ε, διαφωνίες σε σχέση με το κείμενο, αλλά προσβλέπω σε μια καλή και επικοδομητική συνεργασία. Αν Μαρή Μίνα, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη και τους κοιοδησίτες ε, για την έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό και εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα αυτό. Έχουμε εδώ στόχους και απαιτήσει που μερικές φορές ε, έρχονται σε σύγκρουση. Το βλέπουμε καλά και στην έκθεση του κ. Ντόρφμαν. Θέλουμε τον ίδιο, το ίδιο επίπεδο παντού και τιμές ε, προσιτές για τους καταναλωτές και τρόφιμα ύψης της ποιότητας βάσει υψηλότερων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων και τήρηση των στόχων των περιβαλλοντικών και για την κλιματική αλλαγή και μετέχουμε και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών όπου δεν τηρούνται όλοι αυτοί οι κανόνες απαραίτητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τρόπους συναλλαγής βιώσιμους σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα τα τέλη εισαγωγής για τη σόγια και το φινικέλαιο θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να γίνει βιοθανόλη λιγότερο ενδιαφέρουσα. Αυτό θα ήταν σημαντικό για να καταπολεμήσουμε και την αποδάσωση. Θα το συζητήσουμε αύριο νέε ναι, συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών που δεν θα περιλαμβάνουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ε, δημιουργούν τεράστιες βλάβες στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να επηρεάσουμε σημαντικά το τι συμβαίνει όσον αφορά το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε και εμείς δηλαδή να ζητήσουμε εισαγωγικά τέλη για άλλους τύπους ελαίων. Και στον πω επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε στην παραγωγή και την επεξεργασία ως κριτηρία εισαγωγής. Διότι δείτε ποια είναι η κατάσταση του τελικού προϊόντος που έρχεται εδώ διότι δεν γνωρίζουμε καθόλου πώς ε, παράγονται. Έχουμε ε, διάφορες απαιτήσει, ε, αλλά έχουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάτι που επιβάλλουμε στους εισαγωγέ μας εδώ χωρίς να υπάρχει αλλού. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει κάποιο συντονισμός στο διεθνές εμπόριο. όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς. Θεωρούμε ότι για τα προϊόντα διατροφής και για την γεωργία δεν μπορούμε να ε, έχουμε διαφορετικές ε, συνθήκες από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο ή να υπολοιπόμαστε το υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Ζαντό, εκτός μικροφώνου μιλητής. Αλλά για το ζήτημα των χρόνων Μερκουσούρ, όπως γνωρίζετε, ακούγονται πολλά σκάνδαλα υγειονομικά όσον αφορά την κτηνοτραφία βόηου κρέατος και τα σφαγεία στη Βραζιλία. Και ο πρόεδρος Βραζιλίας έμπλεκτε ε, σε ένα σκάνδαλο της εταιρείας GPS που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως ε, βόηου κρέατος δεν αποκλείεται να υπάρχουν κάποιες προθέσεις προστατευτικές αλλά οι Αμερικανοί έχουν μπλοκάρει ε, την εισαγωγή βοήου κρέατος από τη Βραζιλία και εμείς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μαχόμαστε για την προστασία των ζώων του περιβάλλοντος και προσπαθούμε να κρατήσουμε και κάποιους παραγωγούς βοήου κρέατος στην Ευρώπη κάποιους κτηνοτρόφους και θα θέλαμε να μάθουμε πώς έχει λάβει υπόψη τα περιβαλλοντικά προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ξέρετε, η κτηνοτροφία βόηου κρέατος στη Βραζιλία γίνεται ει βάρο του Αμαζονίου με τεράστιο κλιματικό κόστος. Τα προβλήματα υγείας, τι κάνετε για όλα αυτά με όλες αυτές τις συζητήσει που κάνετε, όλα αυτά που λέτε, που τελικά έχουν ως αποτέλεσμα να μην παραμένουν και τόσοι κτηνοτρόφοι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τσάλι παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απαντήσω συνοπτικά στις παρατηρήσεις των μέλων της Επιτροπής για το σχέδιο γνωμοδότησης του κ. Κέλλη. Θα πω και κάποια πράγματα πέραν της έκθεσης. Η Κομισιόν υποστηρίζει τη γνωμοδότηση του κ. Κέλλη. Θεωρούμε ότι γενικά παρουσιάζει κάποια ισορροπία. Σημειώνουμε ωστόσο ότι πολλοί βουλευτές ε, εκφράζουν την άποψη ότι θα έπρεπε να υποθούν περισσότερα για μια πιο βιώσιμη ε, και περιβαλλοντικά ευαίσθητη ΚΑΠ στο μέλλον. Ε, μια κάπου που θα είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς το να συμπεριληφθούν αυτές οι επιθυμίες στην νομοδότηση. Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα προσπαθήσουμε πραγματικά να λάβουμε υπόψη στις πολιτικές ε, τη βιωσιμότητα σε μεγαλύτερο βαθμό την παραγωγή με σεβασμό του περιβάλλοντος, ε, ε, υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και προστασία των ζώων. Το έχω πει. Για να τηρούν αυτά τα πολύ ψηλά περιβαλλοντικά ε, πρότυπα και πρότυπα προστασία των ζώων, όλα αυτά συνεπάγονται πολύ ψηλό κόστο παραγωγή. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό η επόμενη ΚΑΠ να συνεχίσει να παρέχει επαρχή ισοδηματική στήριξη στους ε, αγρότες ώστε να μπορούν να αντιπεξέλθουν σε αυτά τα υψηλά κόστη. Δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, ε, άκουσα ένα-δυο βουλευτέ που αναφέρθηκαν σε ευαίσθητα προϊόντα στο διεθνέ εμπόριο. Συμφωνούμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει τι εμπορικέ μα συμφωνίε μα είναι αδύνατο να απελευθερώσουμε απόλυτα όλα τα γεωργικά προϊόντα. Υπάρχουν κάποιοι ευαίσθητοι τομεί. Αυτό λαμβάνεται υπόψη σε όλε τι διαπραγματεύσει μα. Εξετάζουμε πάντα τι πιθανέ επιπτώσει τη απελευθέρωση σε τομεί όπω το βόλιο κρέο, η ζάχαρη, το Ορίζει οτιδήποτε αναφέρθηκε. Και αυτή η ανησυχία αποτυπώνεται ε, επαρκώς στο σχέδιο ψηφίσματος. Και τρίτον, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ΚΑΠΑ και την ανάπτυξη, η ΚΑΠΑ έχει αλλάξει εντυπωσιακά την τελευταία 20 αιτία. Όπως είπε και ένα μέλος εδώ, δεν επιχορηγούμε πλέον τις εξαγωγές, η εισοδηματική στήριξη προς τους γεωργούς δεν στρεβλώνει το εμπόριο, αναγνωρίζεται από τον ΠΟΕ ότι δεν επιδρά ε, στις ε, τιμές ούτε στην παραγωγή και έχουμε ένα πολύ ανοιχτό εμπορικό καθεστώς με τις ε, χώρες εταίρους. Είμαστε η μεγαλύτερη εισαγωγή μάλιστα προϊόντων που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες με μηδενικούς δασμούς και είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικονομία για τις εξαγωγές των τρίτων των αναπτυσσόμενων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολύ σημαντική ε, αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο ενός σχετικού προγράμματος όπου 62 χώρες ε, δίνουν προτεραιότητα στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιαζόμαστε λοιπόν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια αναπτυξιακής ε, βοήθειας για να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αναπτυσσόμενες ε, χώρες ειδικότερα στην υποσαχάρη Αφρική ώστε οι γεωργοί αυτών των περιοχών να μπορούν πραγματικά να ξεπεράσουν την απλή γεωργία επιβίωσης και να βρουν μια καλύτερη θέση στην ε, αλυσίδα στη διατροφική αλυσίδα αξίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα πέραν του διεθνούς εμπορίου. επειδή η γνωμοδότηση έκανε έκκληση προς την Κομισιόν να υπάρχει συνοχή ε, μεταξύ εμπορικών, αναπτυξιακών και γεωργικών πολιτικών, ε, εμείς αυτό το βρίσκουμε πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δοκλίβα, θέλεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις ιδέες. Θα τις διαβιβάσω στον εισηγητή. Και υπάρχει πάντα αλήθεια σε κάθε άποψη που ακούσαμε. Επομένως, ε, θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ζαντό δεν είναι πολύ ικανοποιημένο γιατί δεν έλαβε απάντηση για το Μερκοσούρ και το πρόβλημα του βόλου κρέατος. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα να κάνω μια απόπειρα να απαντήσω στην παρατήρησή σας. Είναι πάρα πολύ καλή, εύστοχη. Η ουσία είναι ότι με ή χωρίς εμπορική συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εισαγωγές ε, αλλά και η δική μας παραγωγή θα πρέπει να ε, τηρεί τη συγκεκριμένα πρότυπα παραγωγής και ασφάλειας. Εγώ λοιπόν δεν κάνω διάκριση μεταξύ των ε, διαπραγματεύσεων για τη Μερκοσούρ που είναι εν εξελίξη και την εξασφάλιση ότι προστατεύουμε τους καταναλωτές μας στην Ευρώπη εναντίον ε, εισαγωγών που δεν είναι ασφαλείς. Ε, είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και ο ΦΑΟ ε, κάνουν ελέγχους στη Βραζιλία και τα κράτη-μέλη και οι τελωνιακές οι αρχές συνόρων των κρατών μελών εργάζονται πάρα πολύ αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίσουν ότι ό,τι εισάγεται στην Ευρώπη είναι ασφαλές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε και δραστικά μέτρα, αναλογικά όμως, τους τελευταίους μήνες ώστε να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα από τη Βραζιλία ε, που εξάγονται στην Ευρώπη ε, πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ε, αλλιώς δεν μπορούν να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά ούτως ή άλλως. Ωραία. Με αυτό ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 19 Μαρτίου. Συγγνώμη, 27 Μαρτίου, μία η ώρα. Επαναλαμβάνω, 27 Μαρτίου, 1 η ώρα. Θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση 23 και 24 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, περνάμε στο σημείο 7, οι δέσμοι μέτρων για τη στρατηγική δημοσίων προμηθειών. Οι περισσότερες από τις εμπορικές συμφωνίες μας περιλαμβάνουν δημόσιες προμήθειες και φυσικά υπάρχουν και οι συμφωνίες ε, για τις ε, κρατικές προμήθειες. Επομένως ε, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για την ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια επί της επιτροπή για το θέμα αυτό. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και νομοθεσία εν αναμονή, η νομοθεσία IPI, και ο Ντανιέλ Κασπαρή είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης και είναι και ο εισηγητής για την δέσμη μέτρων για τη στρατηγική δημοσίων προμηθειών. Έφτασε και πάνω στην ώρα και του δίνω το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν υπάρχουν ε, ε, έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ του ε, γραφείου, του κτηρίου των γραφείων που έχουμε και της αίθουσα εδώ, είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος την ώρα του. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην γνωμοδότηση για τη στρατηγική δημοσίων προμηθειών, που είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Η έκθεση της ΙΜΚΟ αναφέρει μόνο τη διεθνή διάσταση των δημοσίων προμηθειών σε ένα σημείο. Και επομένω είναι καλή προσθήκη η γνωμοδότησή μα για να τονίσουμε ότι οι δημόσιε προμήθειε έχουν μια σημαντική διεθνή διάσταση και μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικό μοχλό οικονομική ανάπτυξη και θέσεων εργασία στην Ευρώπη λόγω των σημαντικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουμε στον τομέα αυτό. Να, να σας αναφέρω εν συντομία το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Αναφερόμαστε σε πρόσβαση σε τρίτες αγορές, σε διάφανες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις συγκεκριμένε ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον αναφέρει ότι θα πρέπει αφενός να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μέσω ε, πολυμερών συμφωνιών όπως η IPA, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σε διμερείς διαπραγματεύσεις ε, για το εμπόριο τονίζεται επίση η σημασία των δημοσίων προμηθειών όχι μόνο για να υπάρχει πρόσβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξωτερικέ αγορέ, αλλά για να αυξήσουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και να συνάδουν με τα παγκόσμια πρότυπα. Ελπίζουμε μαζί να έχουμε μία σύντομη και ακριβή γνωμοδότηση που θα υπενθυμίσει στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και τη διεθνή διάσταση των δημοσίων προμηθειών. Επίση, θα ήθελα να σα αναφέρω και το χρονοδιάγραμμα προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 10 Απριλίου. Θα τις εξετάσουμε στις 23 και 24 Απριλίου και θα θέλαμε να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση 16 και 17 Μαΐου το οποίο σημαίνει ότι έχουμε άφθονο χρόνο να συνεργαστούμε ε, και να έχουμε καλούς και ισορροπημένους συμβιβασμούς. Θα τη 18 και 19 Ιουνίου στην, Ολομέ... Ε, στην ΙΜΚΟ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν καταρχάς ότι μας έδωσαν ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή και ισορροπημένη γνωμοδότηση και προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία με όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. <laughs> Η Καρολίνα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για, για το σχέδιο γνωμοδότης. Όλοι ξέρουμε ότι η πρόσβαση στις δημόσιες προμήθεια, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και στο τοπικό επίπεδο είναι σημαντική και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών. Έτσι λοιπόν πρέπει και για τι κεντρικέ, αλλά και για τις τοπικές κυβερνήσεις να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο η επιδίωξη μέσα από αυτέ τι προμήθειε των οικολογικών και άλλων προϋποθέσεων ανάπτυξης. Πρέπει να είναι γενικές βέβαια οι διατάξεις. Θα καταθέσουμε κάποιες, κάποιες ε, τροπολογίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Η αρχή της αμοιβαιότητας ε, στην πρόσβαση στις διάφορες αγορές ε, προμηθειών έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας γιατί δεν καλύπτεται πάντοτε υπάρχουν τρίτα κράτη αλλά και εμπορικοί μας εταίροι που προστατεύουν τις αγορές τους από τους Ευρωπαίους υποψηφίους σε πολλές περιπτώσεις προτιμάται η οικονομικά ευνοϊκότερη προσφορά, αλλά εμείς θα θέλαμε πιο οικολογικά, περισσότερα μάλλον ε, οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη για την ε, ε, ανάθεση των προμηθειών. Η επαγγελματοποίηση επίσης ε, των δημοσίων φορέων στις χώρες, η δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιες προμήθειες, σε δημόσιους διαγωνισμούς και αυτών των φορέων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασία, για την ανάπτυξη, για την καινοτομία. Ωστόσο είναι δύσκολη πολλές φορές η πρόσβαση για αυτές σε μεγάλους διαγωνισμούς, σε δημόσιες προμήθειες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό μια μεγάλη ε, σύμβαση να είναι δυνατόν να κατανέμεται σε μικρότερες συμβάσεις ώστε να είναι προσβάσιμες σε αυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης να υπάρχει η δυνατότητα και διασυνοριακής ανάθεσης μέσα από τις δημόσιες προμήθειες. Ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διαφάνεια για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Οπωσδήποτε Χρειάζεται ε, ευχερέστερη δυνατότητα ενημέρωσης και εξασφάλισης πληροφοριών για τις ε, διαδικασίες και τους διαγωνισμούς αυτούς, για τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών και για τις συμβάσεις που συνάπτονται. Βεβαίως εμείς ως ελληνοκράτες θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματική προστασία του πολίτη με μηχανισμούς ε, προστασίας και κυρώσεων. Η ψηφιοποίηση επίσης νέες ψηφιακές τεχνολογίες υπάρχουν, επιτρέπουν και την απλούστευση των διαδικασιών μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Είμαι βέβαια όμω ότι εν τέλει θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή και ισορροπημένη πρόταση. Οι κοινωνικές, οικολογικές, καινοτόμες, δημιουργικές λύσεις θα πρέπει να εμφανιστούν και στις δημόσιες προμήθειες ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ηγεσία μας όσον αφορά τις προμήθειες ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η υλοποίηση ενός ε, καλού πακέτου στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων είναι κλειδί. Υποστηρίζουμε στο ECR την γνωμοδότηση, δημιουργεί ίσες συνθήκες ε, ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι σημαντική πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ωστόσο, τονίζουμε και συμφωνούμε ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί με εταίρους του ΠΟΕ. να διωθεί όλο και περισσότερο σε δημόσιε συμβάσει και να γίνει και διμερό επίση μέσω συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Θέλουμε να δούμε ε, τι ε, να υπάρξει και περισσότερη ψηφιοποίηση στι δημόσιε συμβάσει, να έχουμε ηλεκτρονικέ συμβάσει ε, να γίνουν πιο διαφανείς με αυτόν τον τρόπο οι δημόσιες συμβάσεις, ε, με λιγότερο επαχθείς διαδικασίες και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταπολεμηθούν και οι πρακτικές διαφθοράς ταυτόχρονα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Αυτό θα είναι σημαντικό και για τις επερχόμενες ε, διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Λοιπόν, έτσι, για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συναδελφός μου δεν είναι εδώ, απλά θα διαβάσω τις παρατηρήσεις της. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης για τη στρατηγική δημοσίων συμβάσεων. Η πρωτοβουλία βελτίωσης της υλοποίησης των οδηγιών του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις είναι πολύ επίκαιρη. Όχι μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις εντός της Ένωσης, αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης ε, εμπορικής πολιτικής μας. Όπως ξέρετε, οι δημόσιες συμβάσεις υπερασπίζεται τα συμφέροντα στις, συμφωνίες, ε, στις εμπορικές συμφωνίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόσβαση σε τέτοιες συμφωνίες δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, επηρεάζει σημαντικά και τους φορολογουμένους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες που έχουν τελικά αποκτούν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες χάρη στον ανταγωνισμό. Οι ανοιχτέ αγορέ δημοσίων συμβάσεων είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν όλοι και εμεί και οι εμπορικοί μα εταίροι. Δυστυχώς ε, ε, στην πραγματικότητα πολλές ε, αγορές δημοσίων συμβάσεων σε τρίτες χώρες παραμένουν κλειστές προσφέροντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών δεν εγγυάται σε όλες τις περιπτώσεις πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. ενώ ενθαρρύνει η Κομισιόν τις τρίτες χώρες να συμμετέχουν και αυτές ε, στις, ε, στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να, ε, να, να παροτρύνει η Κομισιόν τις τρίτες χώρες να άρουν τις απαγορευτικές ρήτρε στις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών όσον αφορά την πρόσβαση στις δημοσίες συμβάσεις, να άρουν τα προστατευτικά μέτρα. Ε, κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να αναλύεται περισσότερο η περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων μέσω των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών μας. Τέλος, η ανακοίνωση της Κομισιόν επισημαίνει σημαντικά πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων και αυτό το στοιχείο θα καταστεί σημαντικό. Θα πρέπει να το επισημάνουμε σε σχέση με την εμπορική μας πολιτική, ώστε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους σε αυτές τις αγορές και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τους ε, πράσινους, ο Γιάννη συγγνώμη. Ευχαριστώ. Το βλέπουμε στην περίπτωση του Χάλιβα και της Αμερικής ότι όλο το ζήτημα των βιομηχανικών πολιτικών και των δημοσίων πολιτικών ε, με βιομηχανικούς σκοπούς εντάσσεται σε ένα διεθνή διάλογο και σε έναν ευρωπαϊκό διάλογο. Από πλευρά μου εγώ θα ήθελα σε αυτή την έκθεση να συμπεριλάβουμε και να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει ε, το ε, ενδεχόμενο κάποιες πράξεις ευρωπαϊκής οι εμπορικοί μα εταίροι χρησιμοποιούν τέτοιου είδου εργαλεία για να ευνοούν κάποιους στρατηγικού τομείς, για να προστατεύουν ε, κάποιες επενδύσεις που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίε και για την οικονομική μας εθνική κυριαρχία. Ε, εκ μέρου των Πρασίνων λοιπόν έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις ε, τροπολογιών όχι για να συμπεριλάβουμε σήμερα μια τέτοια πράξη στην νομοθεσία, αλλά για να διερευνήσουμε τη σκοπιμότητα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτού του είδου το μέσο για άλλη μια φορά και για να καταλήξουμε να έχουμε ένα επίπεδο θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορών χωρών. δεύτερων, όπως ε, κάναμε και με τον σύντροφο Φέλνερ, ο οποίος έγινε λόγο, τον απασχολούν ειδικότερα, ιδιαίτερα τα κοινωνικά δικαιώματα παγκοσμίω. Όπως το λέει μόνιμα στο σουηδική σκηνή ζήτω το περιβάλλον, ζήτω η κοινωνία, ζήτω η κοινωνική διάσταση. Και όπως κάναμε, γράψαμε και στην εκθέση Τσίκου, έχουμε συμπεριλάβει τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα η νομοθεσία μας σε όλες τις διατάξεις anti-dumping. Δεδομένων των φιλοδοξιών της Ευρώπης όσον αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού και δεδομένου το ότι θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμητο ανταγωνισμό και στις δημόσιες συμβάσει, πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να εντάξουμε με παρόμοια γλώσσα, όπως αυτή που χρησιμοποίησαμε στην έκθεση Φιάλινα και Τσίκου, το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών συμφωνιών και ειδικότερα την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέλμιν Σόλτς για την ΚΟΕ. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον Ντάνιελ Κασπάρη, τον εισηγητή μας, για την κατάθεση της ε, γνωμοδότησης και την ε, ιδιαίτερη μέρημνα να μην ξεφύγει από τον τομέα της, ε, του εξωτερικού εμπορίου. Στις δημόσιες προμήθειες, ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι εμείς βλέπουμε ως ομάδα πολύ περισσότερα πράγματα από τη μια αγορά για τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να παραπέμψω στα λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανακοίνωσή της και παραθέτω. Οι Ευρωπαίοι πολίτες από την χρήση του χρήματος που συλλέγεται από τους φόρους τους περιμένουν μια πολύ πιο αποδοτική χρήση ε, και υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν καλές ε, επενδύσεις ε, σε πόλεις ευφυείς, ε, όπου μπορεί κανείς να ζει καλύτερα με ασφαλείς δρόμους, με πλατείες, με πάρκα για παιχνίδι, ασφαλείς υποδομές υψηλής ποιότητας, νοσοκομεία με ε, ευχερή πρόσβαση και μέρημνα για τους ασθενείς, με κατάλληλο νοσοκομιακό εξοπλισμό και με τις πιο ε, προωθημένες, με, τις με τα καλύτερα τεχνολογικά ε, Αυτό δηλαδή τι μας λέει. Μας λέει ότι θέλουμε όχι το φθηνότερο αλλά το καλύτερο. Ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα πράγματα σε βιωσιμότητα, σε επενδύσεις, με αποδοτικότητα, σε βελτίωση των όρων ζωής. Και γι' αυτό η δική μας γνωμοδότηση πιστεύουμε ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να τονίζει ότι οι δημόσια αυτές προμήθειες θα πρέπει να επιδιώκουν την ε, υλοποίηση των δικών μας απαιτήσεων ποιότητας, να προσφέρουν δυνατότητες για απασχόληση και να μεριμνούν ώστε να μην ε, γίνεται η επιλογή για την ε, κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου μόνο με βάση την ε, επιλογή ενός ή του πιο φθηνού κατά το δυνατόν δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα ο πληθυσμό μένει άνεργος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια προγραμματική προσέγγιση για να είναι σωστή η χρήση των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Πρέπει σε αυτό μέσα από έναν ε, ε, μέσα από μια δέσμευση ρητή σε όρους συγκεκριμένους να το ε, επιδιώξουμε και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις προτάσεις που κάνει ο συγητής μέσα στη γνωμοδότηση τις σχετικές με την ΠΟΕ και θα αναφέρω τα εξής από την ΠΟΕ ότι η Κίνα λοιπόν μας λέει ΠΟΕ Ε, λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή, ο ΠΟΕ για την ε, Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη δυνατότητα για υπέρβαση το εξές ε, των όρων προσφοράς για τις δημόσιες προμήθειες. Ε, εν περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε και οι δικές μας τροπολογίες θα είναι επικοδομητικές με ιδιαίτερη έμφαση στις δικές μας προτάσεις. Ο κύριος Δάτνχαους. Πρόεδρε, με χαρά βλέπω στο πιδάλιο τον αγαπητό φίλο Ντανιέλ Κάσπαρη και πάλι και είναι μόνο και μια γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία στο επόμενο δεκάμινο. Ε, καταρχάς, Στην ημερήσια διάταξη βλέπουμε τον όρο δημόσιε προμηθείε. Α, τι ωραία, θα πει κανεί. Πάω πάρω καφέ καλύτερα γιατί βαριέμαι. Και όμω όχι, γιατί η πρώτη ρήτρα αυτή την, ε, σε αυτό το πρώτο εδάφιο, σε αυτή τη γνωμοδότη στο σχέδιο, μα λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι δημόσιε προμήθειε είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα μα απασχολήσουν στο, κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Όταν ήμουν υποψήφιο, πάλι ποτέ, το 1974, εκ μέρου του Συντηρητικού Κόμματο, ε, υποψήφιο βουλευτή, ε, έβλεπα ότι ο κόσμο έλεγε πάντα θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ανοιχτέ ε, δημόσιου διαγωνισμού με διαφάνεια και που να μην αποκλείουν κανέναν. Βλέπουμε βεβαίω το σημαντικό όφελος το αξιόπιστο, βαθύ όφελος του να έχουμε διαφάνεια, το να έχουμε διαγωνισμούς χωρίς αποκλήσεις. Και βεβαίω τώρα μην δίνονται με απευθεία ανάθεση δημοσίες δημόσιε σε κάποιο φίλο, ε, ωστόσο, και εδώ δεν έχω απάντηση, υπάρχει το εξή. Δεν θα πρέπει να ευνοούνται οι ε, ντόπιοι, οι εγχώροι ε, έναντι κάποιων ε, που θα έρθουν από έξω να ζητήσουν μια δημόσια σύμβαση στην Νοτιοανατολική Αγγλία, από την οποία εγώ εκλέγομαι και που έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή τροφίμων. Δεν θα έπρεπε να προτιμούνται φερρυπίν για τα γεύματα των σχολείων ή τοπικές επιχειρήσεις. Και όμως αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι λοιπόν αυτό και βεβαίως ε, το επισημένο και ο συνάδελφος και αγαπητός ε, αντιπρόεδρος κ. Αντώ το είπε ήδη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα. Και με τον κύριο Σόλτ πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά επίσης πολλές φορές συμφωνούμε, πράγμα το οποίο μπορεί να ξαφνιάζει κάπως. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δεν είμαστε υπέρ της ε, πολιτικοποίησης του εμπορίου, ούτε είμαστε κατά της πολιτικοποίησης των ε, δημοσίων προμηθειών. Ωστόσο δεν θα πρέπει οι δημόσιες προμήθειες να χρησιμοποιούνται ε, σαν ε, παραθυράκι μέσα από το οποίο θα περάσουν πολιτικές επιλογές που δεν μπορούν μέσα από την ανοιχτή πόρτα ή θύρα να περάσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόσωπος της ε, Με χαρά ακούμε τόσο πολλά κολακευτικά λόγια για το ε, δέσμη αυτών μέτρων εθελοντικής φύσεως για τις δημόσιες προμήθειες. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σαφή θέση και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και τις ε, αρχές ε, που συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις ε, να ε, αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες προμήθειες με πιο στρατηγικό τρόπο. Ο λόγος είναι ότι το 40% του ΑΕΠ της Ευρώπης δαπανάται για δημόσιες προμήθειες, που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για να έχουμε όχι μόνο καλύτερη αξία για τα χρήματα που δαπανούμε, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε ως στρατηγικό ε, στόχο για ευρύτερους στόχους, για παράδειγμα μια οικονομία χαμηλότερη σε χρήση άνθρακα, πιο δίκη κοινωνία και καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Αναγνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός εξακολουθεί ε, να είναι ε, ουσιαστικό στοιχείο των δημοσίων προμηθειών, θεμητή πρόσβαση και βελτιωμένη πρόσβαση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά επίση, ενθαρρύνουμε τι δημόσιε αρχέ να εξετάσουν και την ευρύτερη καλύτερη ένταξη και άλλων στοιχείων και όχι μόνο τη χαμηλότερη ε, τιμή. Να υπάρχουν και ποιοτικά κριτήρια τα οποία ε, σε εξυπηρετούν και ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όσον αφορά τις διεθνείς διαστάσεις, ε, ε η καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες προμήθειες και ε, εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρχουν καλύτερες, περισσότερες δημοσιεύσεις, να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα υποβάλουν προσφορά ώστε να μπορούν ε, να συμμετέχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δημόσιες προμήθειες, αλλά να εφαρμόσουμε την ίδια φιλοσοφία και εξωτερικά σε διεθνείς αγορές. Ο αυξημένο ανταγωνισμός, οι ανοιχτές αγορές, ε, κατά την άποψή μα είναι η άγουσα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε ε, μέσω ε, προβολών των προτύπων μας σε δημόσιες προμήθειε και στο εξωτερικό, σε χώρες στι οποίε υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των ίδιων προτύπων και ανοιχτό πνεύμα. Υπάρχει και μια ομάδα στο GPA που περιλαμβάνει στοιχεία διαφάνεια για το πώ μπορούμε να συλλέγουμε καλύτερα δεδομένα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και μέσω πιο φιλόδοξων διμερών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Όλοι ζητάμε μεγαλύτερη φιλοδοξία σε αυτές τις συμφωνίες. Αναγνωρίζουμε ότι ε, η αμοιβαιότητα δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη όσο θα επιθυμούσαμε και ε, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει κάτι το οποίο περιλαμβανόταν και στην προηγούμενη ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την προώθηση της παγκοσμιοποίηση. Ε, χρειαζόμαστε διαφορετικά μέσα και εργαλεία και ζητάμε και από τους συνομοθέτε να επιταχύνουν τι εργασίε για το μέσο IPI. Αλλά εν τέλει αυτό το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αν παραμείνουμε ανοιχτοί και αν δεν υποκύψουμε στο προστατευτικό κλίμα των άλλων χωρών, θα συνεχίσουμε να έχουμε ε, έναν άσο στο μανίκι μας. Ε, φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες από πουδήποτε, από το Κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη, όσον αφορά ε, πιο δραστήρια μέτρα ή έστω και μια νομοθετική πράξη για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά προϊόντα και φυσικά είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συζήτηση. Πιστεύουμε ότι ο ανοιχτό ε, ανταγωνισμός είναι στο επίκεντρο των δημοσίων προμηθειών και σε εσωτερικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο και επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας ώστε το επίπεδο φιλοδοξίας των δημοσίων προμηθειών και της διαφάνειας να προχωρήσει περαιτέρω ε, και στις διμερείς ε, συμφωνίες εμπορίου αλλά και ε, σε πολυμερείς συμφωνίες. Είναι αλήθεια ότι ε, όλοι όσοι κάνουν αίτηση δεν παρουσιάζουν παρκώς φιλόδοξες προτάσεις ε, στο GPA, αλλά συνεργαζόμαστε και με άλλες πλευρές ε, για να ζητούμε και να διαπραγματευτούμε καλύτερες προτάσεις και παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ο Ντανιέλ Κασπαρή. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. από ό,τι αντιλαμβάνουμε κάποια πράγματα είναι αντίστροφα. Για παράδειγμα, είναι ο συνασπισμό μετά, μεταξύ του Γιάννη και του Ντάτμα, το γεγονός ότι υπερασπίζεστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα εμπορίου, αλλά είμαι βέβαιος ε, ότι μετά την ε, κατάθεση των τροπολογιών τα πράγματα θα ξανάρθουν στη θέση τους και προσβλέπω σε καλούς ε, συμβιβασμούς και να έχουμε μια καλή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ωραία. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Τρίτη 10 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Με αυτό ολοκληρώνεται και το σημείο 7 και τώρα πάμε στο σημείο 8 το οποίο είναι και κλεισμένο των θυρών. Θα διακόψουμε για ένα λεπτό λοιπόν. Όποιος δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην αίθουσα στα μέλη βεβαίως η Επιτροπή, η Γραμματεία, η ε, Νομική Υπηρεσία, η Πολιτική Ομάδα, η Βοηθή μπορούν να παραμείνουν. Οι υπόλοιποι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα και μάλιστα γρήγορα.